επόμενο θέμα συζητήσει για περιπτώσει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Το πρώτο θέμα είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κρυμαία, ιδίω των Τατάρων τη Κρυμαία. Uh, Άρχεται η συζήτηση. Θα δώσω μέσα στο λόγο στου συντάκτε. Πρώτο ο κύριο Μπιτζικόφερ για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο και επίκαιρο το Κοινοβούλιο σε ένα κοινό ψήφισμά του να τονίσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην κατεχόμενη Κρυμαία, στα κατεχόμενα εδάφη της Κρυμαίας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Τατάρους της Κρυμαίας, οι οποίοι υφίστανται διώξεις από την αρχή ακόμα την ίδια της ρωσικής εισβολής. Οι εκλεγμένοι τους εκπρόσωποι δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με βάση την ετολή τους, τους απαγορεύεται αυτό, uh, όπως κανονικά θα έπρεπε να κάνουν σύμφωνα με τον Ουκρανικό νόμο. Τι έκανε η Ρωσία και τι συνεχίζει. Καταστολή των Τατάρων της Κρυμαίας, διότι είναι ευρύτατη η καχυποψία και η δυσπιστία που έχει η Ρωσία απέναντι σε αυτό τον πληθυσμό. Πιστεύουμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη του και με χαρά ε, έχουμε καταθέσει το κοινό αυτό ψήφισμα. Ευχαριστώ. Κυρία Φωτήκα, ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν από δύο χρόνια, Πρόεδρε, είχαμε μία πολυεθνική Ε, και είχαμε μια ομάδα από βουλευτές από πολλά έννοια και μαζί με την κυρία Μογκερίνη πήγανε επί Γιαννουκόβης τότε ε, στη ε, Κίεβο το επανάσταση του Αϊντάν θα γινόταν σε λίγες μέρες τότε. και μετά από κάποιες εβδομάδες είχαμε την, την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας και θυμάμαι ότι πήγα τότε εκεί και κοίταξα αυτά τα πρόσωπα του, του κόσμου και που μου δείξανε από πού οι ελεύθεροι σκοπευτές ε, σκότωσαν τον κόσμο. Μίλησα ε, σε πάρα πολλούς ε, Ουκρανούς και μου είπαν ότι αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος είναι η, την αλλαγή παρά όλες τις δυσκολίες. Οπότε χρειάζεται αλληλεγγύη και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, κατάληψη της Κρυμαίας. Δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί η παράνομη προσάρτηση και θα πρέπει επίσης να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο που να μην μειωθεί η ελληνική μας. Ε, θα επιδείξουμε δυναμία να αλλάξουμε την ε, στρατηγική μας, οπότε θα πρέπει όλοι να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο. Παντσέρι, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι έχουν ενταθεί οι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη ε, προσάρτηση από τη Ρωσία τη Κρυμαία και έχουμε διάφορου ε, διεθνεί ε, φορεί που έχουν αναφέρει σχετικώ όλα αυτά που γίνονται κατά τη κοινότητα των Τατάρων, γιατί περισσότερο από του Τάταρου θα είναι κατά τη προσάρτηση και επίση σαμποτάρανε το Δήμο τη 15η Μαρτίου και επίση είδαμε ότι τώρα έχουμε άσκηση βία, έχουμε βασανισμούς και ε, έχουμε παράνομες δίκες. Είδαμε τι γίνεται τώρα με την ε, απονομή της ρωσικής ε, ηθαγένειας που όποιος δεν την έχει υφίσταται αυτές τις διακρίσεις οπότε θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι το τι έχει γίνει με τους δημοσιογράφους που φεύγουν από την Κρυμαία γιατί υφίστανται διώξεις. Άρα θα πρέπει εγκριθεί ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Πρέντεν, επόμενο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους σήμερα συζητούμε την κατάσταση της Κρυμαίας. Η πολιτική μου ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, προσπαθεί ένα εξάμεινο και πλέον να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτηση για την Κρυμαία. Και πρέπει να πω ότι άλλε πολιτικές ομάδες αντιτάχθηκαν σε αυτό. Οι μόνοι που μας υποστήριξαν ήταν οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Ε, από την αρχή και μέχρι ε, τώρα. Για ποιο λόγο. Έχουμε μια επαμφωτερή στάση απέναντι στην ε, Ρωσία και την Κρυμαία. Μια μεγάλη σημαντική πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο μα ζητάει να μεταβούμε σε επίσημη αντιπροσωπεία στη Μόσχα. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα πιστεύω. Όσο όλοι οι συνάδελφοί μας ε, της ε, Βουλής που βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Κρεμλίνου δεν έχουν ε, αφαιρεθεί από τη λίστα αυτή και, όσο συνεχίζει να κατέχει τα εδάφη της Κρυμαίας η Ρωσία δεν μπορούμε να έχουμε εξομάλυνση σχέσεων. Ευχαριστώ. Γκοζάλια Ρισπένια, σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Κρυμαία τι βλέπουμε. Πώς τα γεωπολιτικά συμφέροντα έρχονται αντιμέτωπα με τη ζωή του πληθυσμού. Μας ανησυχεί η κατάσταση του κόσμου. Αυτό δεν θα λυθεί ούτε με τον αποκλεισμό και τον εμπάργο. Ε, υπάρχει ένα δράμα εκεί που ζει ο άμαχος πληθυσμός. Και αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάσταση ε, των Τατάρων και άλλων μειονοτήτων, εθνικών μειονοτήτων. Οι εθνικέ μειονότητε και οι αυτόχθονοι πληθυσμοί έχουν δικαιώματα που θα πρέπει να γίνονται σεβαστά παντού στον κόσμο και στην Κρυμαία. Για όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται ε, διαπραγμάτευση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ε, όροι και προϋποθέσεις για να μπουν δημοσιογράφοι, ανθρωπιστική βοήθεια και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε ε, σε όλη τη διάρκεια επίλυση αυτή τη διαφορά. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής ε, των ε, συντακτών, ο κύριος Οστριβίτσιος. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρο τη Ρωσίας, η τελευταία του συνέντευξη στην είπε οι νασιολιστικές ομάδες στην πρωτεύουσα στο Κίεβο ε, σκότωσαν ανθρώπους στην Κρυμαία. Και τι να κάνουμε, να μην πάμε εμείς σε πόλεμο, εφόσον είχαν σκοτωθεί άνθρωποι. Ναι, αλλά συμπεριφέρεται σαν ε, επιτελής. Είναι όμως δικιά σας ευθύνη κύριε Πούτιν, οι αγνοούμενοι ή οι δολοφονημένοι από το 2014 στην Κρυμαία. Οι Τάρταροι που έχασαν τη ζωή τους είναι δικιά σας ευθύνη. Ο Τζαβούρ, ο Τάρθοφ, ο Ζενεντίνοφ, ο Ισλάμ Τζιπάροφ, ο Τζεφτέφ Ισλάμοφ, ο Σκαντέρα Ψαλάμοφ, ο Ρουσλάν Κενίερ, ο Ριλέν Τερέκοφ και ο κατάλογος δεν είναι πλήρης βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι. Μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του 20ου αιώνα. Ας ονομάσουμε τα πράγματα με το πραγματικό τους όνομα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Τώρα ο πρώτος ομιλητής ο κύριος Πλένκοβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ψήφισμά μας στηρίζει την ελεύθερη επιλογή της Ουκρανίας να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πορεία και επιστένει την προσοχή τη διεθνού κοινότητα, στις σοβαρέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την παράνομη κατάληψη από τη Ρωσία. Η Τάρταρη, που είναι αυτόχθον ο πληθυσμό, υποφέρει από καταχρήσει και από τη ε, συμπεριφορά των αρχών εκεί. Πρέπει να παραμείνουν οι κυρώσει σε βάρο τη Ρωσία. Αν οι ρωσικέ αρχέ θέλουν να βελτιώσουν τι σχέσει του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να αποσυρθούν από την Κρυμαία και να επιτρέψει την Ουκρανία να διαχειριστεί τα εδάφη τη. Οι διεθνεί οργανώσει, μη κυβερνητικέ οργανώσει, τα μέσα ενημέρωση πρέπει να έχουν πρόσβαση στην Κρυμαία και να υπάρχει συντονισμό με τι Ουκρανικέ αρχέ. Γι' αυτό και καλωσορίζω την επίσκεψη του δικού πεσταλμένου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στηρίζω επίσης και την ε, πρόταση για μια Γενέβη ΣΥΝ. Η Κρυμαία πρέπει να επιστρέψει στην Ουκρανία, να σταματήσει η κατοχή στα Ανατολικά και γνωρίζουμε ότι η αιτία των προβλημάτων εκεί είναι μία και μόνο. Ευχαριστώ κύριο Σάνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις εδώ μέσα θέλουν να λυθεί το πρόβλημα στην Κρυμαία. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα ποιο είναι είναι να σταματήσουν αυτές οι θηριωδίες του Πούτιν κατά των ε, κατοίκων της Κρυμαίας. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μειονότητα των Τατάρων αναφέρομαι. Καταβάλουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχουν και απόπειρες ε, υπονόμευσης της αλληλεγγύης. Και αυτό είναι δώρο στον Πούτιν. Οτιδήποτε λοιπόν μας υπονομεύει και ε, μας διχάζει ε, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Πούτιν. Καλό λοιπόν όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ε, προσιλωμένοι στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να μην υπονομεύουμε την ίδια μας την πολιτική για κάποιους απότερους σκοπούς και με ιστεροβούλια. Ο κύριος Ντεμές Μάρκερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όποιο έχει επισκεφτεί την Κρυμαία σε καλύτερου καιρού γνωρίζει ότι ε, ήταν πολύ ζωντανό ο τουρισμό. Ήταν αψηφιωτό, ωραίο, διαφόρων γλωσσών, πολιτισμών και παραδόσεων. Εγώ έκανα ένα γύρο λίγου μήνε πριν ε, την προσαρτήση Ρωσία. Ένα κόσμημα ήταν ε, στη Μαύρη Θάλασσα και τώρα είναι η χερσόνησο του φόβου. Από την παράνομη προσάρτηση ακολουθεί η Ρωσία του Πούτιν μεθόδου χωρί καμία τύψη. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι λένε οι αρχές. Είτε σας αρέσει αυτά που κάνουμε, να σας αρέσουν ε, ε, να ε, κλείσετε το στόμα σας, αλλιώς να φύγετε. Διώκονται οι Τάταροι, οι δημοσιογράφοι, οι ακτιβιστές είναι παράνομοι. Οι Τάταροι είναι θύματα απαγωγών, δολοφονιών και βασανιστήριων. Επαναλαμβάνεται η ιστορία για αυτό τον περήφανο λαό. Είναι έσχο. Επιτέλου, έφτασε η αποστολή του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Θα πρέπει η Ρωσία να συμμετέχει και στι τελικέ ε, ε, φάσει και στα τελικά συμπεράσματα τη έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Κάλλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο λόγος για τους οποίους ε, καταστέλει την ελευθερία έκφρασης και σκέψης η Ρωσική Ομοσπονδία σε αυτή την περιοχή είναι ακριβώς ε, διότι υπάρχουν σοβαρές επικρίσεις σε αυτή την περιοχή κατά της Ρωσίας. Είναι ακτιβιστές ε, οι Τατάροι και είχαν ε, υπερασπιστεί τη σημαία της Ουκρανίας σε μαζικά συλλαλητήρια ήδη από το 1900 από την ίδρυση της Ουκρανίας ήδη από το 44 είχαν εξεγερθεί ε, κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ε, και ε, τώρα όσοι δεν δέχονται την ρωσική υπηκότητα δεν μπορούν να έχουν για τα παιδιά τους θέσεις στα σχολεία, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Διώκονται λοιπόν οι Τατάροι και παραβιάζονται όχι μόνο ανθρώπινα δικαιώματα αλλά τίθεται εν κινδύνο συγγνώμη, η γλώσσα τους και ο πολιτισμός τους. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Ε, και να μιλάνε τη γλώσσα τους. Ευχαριστούμε κύριο Στέπινα ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το δικαίωμα των ε, Τατάρων για εκπαίδευση στην γλώσσα τους δεν γίνεται σεβαστό. Ο αριθμός των σχολείων που διδάσκουν στην Ταταρική μειώνεται, κάποια σχολεία κλείνουν δια της βίας συμβολικά και πολιτιστικά στοιχεία της ε, ταταρικής ταυτότητας ε, καταστέλλονται. Και οι ηγέτες τους ε, διώκονται. Ο Μουσταφά Τζαμίλιεφ εδώ και καιρό έλεγε πως η Ρωσία ήθελε να καταλάβει την Κρυμαία. Ο δε κύριος Τζαμίλιεφ το 1968 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση στην Έσεσοδο επειδή καταδίκασε την ε, κατοχή της δικής μου χώρας τότε, της ε, Τσεχοσλοβακίας. Καταδικάζονται δε με κάτι απίθανα άρθρα του ρωσικού ποινικού κώδικα, ενώ ε, θεωρητικά η Κρυμαία είναι ακόμα έδαφος της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ. Τα δύο εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στην Κρυμαία αντιμετωπίζουν φοβερές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ταταρική κοινότητα όπως και για όσους άλλους αντιστάθηκαν στην παράνομη κατοχή και προσάρτηση της ε, Κρυμαίας. Το αποτέλεσμα είναι απαγωγές, βίαιη καταστολή και τα λοιπά. Και σημαίνει επίσης πως δεν υπάρχει πρόσβαση σε διεθνείς φορείς στου οποίου μπορούν να στραφούν οι Ευρωπαίοι όταν ε, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό της ε, κοινότητας των Τατάρων της Κρυμαίας καθώς και στο πλευρό όλων των Ουκρανών που θέλουν να διατηρήσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους. Καλό την Ρωσική Ομοσπονδία και τις de facto αρχές στην Κρυμαία να αφήσουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς. Ο κ. και ένα λεπτό. Πρόεδρε, μετά την βίαιη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία το 2014, ο πληθυσμός των Τατάρων της Χρυσονήσου και η Ρώσικη μειονότητα έχουν υποφέρει υποβάθμιση των βασικών τους ελευθεριών και δικαιωμάτων. Οι Τάταροι έχουν μποκοταριστεί από το ε, ψεύτικο, το ψευδές δημοψήφισμα για την ε, κυριαρχία της Ρωσίας και έχουν επανέλθει στο πρόγραμμα του Στάλιν και της Μόσχας για την ε, εξορία τους, όπως γινόταν τη δεκαετία του 40. Καταστέλλονται οι ελευθερίες τους και οι δημόσιες εκδηλώσεις τους έχουν απαγορευτεί. Οι συλλήψεις έχουν γίνει πια κοινότοπο φαινόμενο στην Χερσόνησο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ ενισχυτικά. Καταδικάζω λοιπόν ε, την ε, προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία που ήταν μέρος της Ουκρανίας και καλώ τις αρχές να σεβαστούν το περιεχόμενο των βασικών ελευθεριών των και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις τους με τους Τάταρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τους παρακολουθεί πολύ προσεκτικά. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ο κύριος Συναδεινός. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση άγεται και φέρεται και έχει καταντήσει να εκφράζει τη γνώμη μόνο συγκεκριμένων χωρών και κέντρων εξουσίας και ειδικά της γερμανίας. αν μη τι άλλο είμαστε υποκριτές όταν συζητάμε για τους περιορισμούς των θρησκευτικών δραστηριοτήτων στην κρυμαία τη στιγμή που η αγία σοφιά αν και αποτελεί ναό ορθόδοξης χριστιανικής της πίστεως απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως λαδευτικό τόπος των χριστιανών από την τουρκία που επιδιώκει να γίνει μέλος της ένωσης. μιλάτε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τι δυνάμει κατοχή στην κρυμαία. πότε έγινε η εισβολή και από ποιον στην κρυμαία; δεν μα είπε ο εισηγητής ταυτόχρονα κάνετε τα στραβά μάτια για τις αθλειότητες των τουρκικών δυνάμεων κατοχής στην κύπρο. πολιτική διαστροφή θα χαρακτηρίσω το να θέλετε την τουρκία να σας εφοδιάζει με τζιχαντιστές με ισλαμικούς εξτρεμιστές με λαθρομετανάστες και με ναρκωτικά από τη μέση ανατολή γιατί αλλιώς δεν εξηγείται η οποία με τον νεοοθωμανισμό και το δόγμα του στρατηγικού βάθους ενδιαφέρεται για τη μειονότητα του 12% των τατάρων τους οποίους εδώ και 20 χρόνια τροφοδοτεί και εφοδιάζει και σα οδηγεί στη σύγκρουση με τη ρωσία. Αποφέγετε τη σύγκρουση με τη ρωσία βρείτε κοινό τόπο συμφερόντων και προσπαθήστε να ομαλοποιήσετε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή τη Ευρώπη. ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. μια δικασία Διαδικασία Κατσδιάη. Μακροσκέλης κατάλογος, έχω μόνο δύο λεπτά, οπότε θα επιτρέψω μόνο σε δύο αγορητές, ο κύριος Πόσπιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να σχολιάσω αυτό που μας είπε και ο κύριος Στέτιν. Είμαι Τσέχος και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Μουσταφέ Τζαμίλη διαδήλωσε κατά ε, της ε, Τσεχοσλοβακίας ε, και μπόρεσε να υποστηρίξει αυτή τη χώρα που καταπιέστηκε από την Σοβιετική Ένωση καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυτό συμβαίνει τώρα και στην Κρυμαία. Θα πρέπει να σταματήσουμε τον εκφοβισμό των Τατάρων και να φροντίσουμε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα τους. Ε, έψιλον εκφοβισμοί, απαγωγές, εξαφανίσεις επίσης 20.000 ε, τάτερ φύγανε από την ε, Κρυμαία λόγω ε, της καταπίεσης τους και προσπαθούν να πάνε στην Ουκρανία. Πάλι πρέπει να φύγουν από τα πάτρια εδάφη τους, θα πρέπει να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία. Εγώ σε κάθε λομέλη σχολιάζω αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Σήμερα στο Στρασβούργο μιλάμε και ακούγεται η φωνή των Τάταρων της Κρυμαίας. Η κατάσταση εκεί πέρα είναι συνέπεια της ε, προσάρτησης τους από την ε, Ρωσία. Δεν μιλάμε όμως για τις δικές μας αποφάσεις. Χτες ε, μάθαμε για το τι έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν ακούσαμε τίποτα. Κιχ για την Κρυμαία, τις συμφωνίες του Μίνσκ και την πολύ σοβαρή απειλή των επιθετικών βημάτων που μπορεί να λάβει η Ρωσία και οι φιλορωσικές δυνάμεις. Τέλος, δεν ακούσαμε τίποτα για τον Nord Stream 2. Το έργο αυτό τελικά καταλήγει στο τίποτα και αναστρέφει τα αποτελέσματα των κυρώσεών μας στη Ρωσία. Δεν αντιδρούμε όσο στεναρά θα έπρεπε. Και δεν αντιδρούμε και που θα έπρεπε. Έχετε κάτι επί της διαδικασίας να πείτε. Κύριε Μπιουτικόφερ, κυρία Πρόεδρε, ζήτησα να αντιδράσω σε μια προσωπική επίθεση. Και θα ήθελα να σημειωθεί παρακαλώ στα πρακτικά στις ε, παρατηρήσεις μου. Είπα πως ήταν θετικό ότι έξι πολιτικές ε, ομάδες κατέληξαν σε κοινό ψήφισμα και η συζήτηση κατέληξε ότι είμαστε ενωμένοι. Λυπούμε άρα για το ότι ο κύριος Πρέντα ε, χρησιμοποίησε τον χρόνο ομιλίας που είχε ως συντάκτης να επιτεθεί σε άλλους συναδέλφους και σε μένα και είπε ότι όσοι δεν στήριζαν τις προτάσεις του ΕΛΚ νωρίτερα δείχνουν μια στάση επαμφωτερίζουσα απέναντι στην ρωσική κατοχή της Κρυμαίας. Είναι αναλυθές αυτό, άδικο, διχαστικό και απορρίπτω αυτή την κατηγορία. Ευχαριστώ. Το σημειώνουμε λοιπόν με βάση το άρθρο 164. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης από την ρωσική Ομοσπονδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εξακολουθεί να καταγγέλει αυτό το περιστατικό και εξακολουθεί να μην το αναγνωρίζει. Κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πέραν αυτού έχει και σοβαρότερε επιπτώσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παράνομη προστάτες Κρυμαία, ε, συστηματική παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατοίκων της Κρυμαίας, ε, βασική παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών σε αυτή την Χερσόνησο και επιβάλλεται η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ε, και επικρατεί νομική ανασφάλεια και διακριτική μεταχείριση. Η κοινότητα των Τατάρων ε, και άλλοι κάτοικοι που υποστηρίζουν την εδαφική ακαιρεότητα της Κρυμαίας ε, καταβάλουν πολύ ακριβό τίμημα για τις απόψεις τους. Στη Συμφερούπολη, παραδείγματο χάρη, για την απέλαση για την, του 1994 δεν επιτράπηκαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο ε, και οι ακτιβιστές ε, Τατάρι διώκονται ποινικά. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές εκκρεμείς υποθέσεις εξαφανίσεων, βασανιστήριων και δολοφονιών νέων Τατάρων οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί καν από την αστυνομία. Η κυρία Μογκερίνη συζήτησε το ζήτημα όταν προσωπικά συναντήθηκε με εκπροσώπους των Τατάρων στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2015. Θα ήθελα επίσης ε, να τονίσω τα περί κράτησης ε, ε, και ποινών φυλάκισης των των Τατάρων ζητούμε την άμεση αποφυλάκησή τους και την ασφαλή επιστροφή τους στην Κρυμαία. Ε, επίσης ε, θέλουμε σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας ε, συμπεριλαμβανομένης και της Συμφερούπολης να επάψει άμεσα η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέρα από την απελευθέρωση των Σέντσοφ και Κολσένκο και υπάρχουν τον Την άνοιξη το 2015 έγιναν ανεπίσημες επισκέψεις, διαρκώς ε, δραστηριοποιούνται οι αποστολές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, από εκπροσώπους των Τατάρων εντός και, εκτός, εντός και εκτός συγγνώμη, της Κρυμαίας ε, και έχουμε τεκμήρια σε σχέση με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρησιμοποιούμε πολυάριθμες πηγές και ελπίζουμε ότι με την τελευταία επίσκεψη ε, του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, υπό την αιγίδα του ε, στρατηγού Στούτσμαν θα μπορέσει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην Κρυμαία. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχω λάβει 7 διαφορετικά ψηφίσματα, προτάσεις ψηφίσματος για αυτή τη